στην ε, ομάδα στην οποία προεδρεύω, στο Financial Assistance Working Group και εμείς ε, τοποθετηθήκαμε σχετικά με την ελληνική υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερικής διάταξης που έχει να κάνει με την έκθεση της κυρίας Πιετικάινεν. Ευρωπαϊκές Εταιρείες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή οικονομία εξαρτάται πάρα πολύ από τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Κλάδο και φυσικά αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει να κάνει και με την ε, χρηματοδότηση. Η απόκτηση χρηματοδότηση αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, το θέμα αυτό, χρειαζόμαστε καινοτόμου τρόπου χρηματοδότηση ε, για επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου και μιλάμε και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για πιο μεγάλα έργα. Χρειαζόμαστε πιο πολύ κεφάλαιο επιχειρηματικότητας Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο πολλά επιχειρηματικά κεφάλαια. Απέχουμε πάρα πολύ από το σύστημα α, των ΙΠΑ, όπου το επιχειρηματικό κεφάλαιο είναι πενταπλάσιο σε όγκο. Και φυσικά όλα αυτά οργανώνονται σε εθνικό επίπεδο. Αυτό περιορίζει φυσικά την ε, δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό σε περιοχές ε, και κλάδους όπως είναι αυτός του περιβάλλοντος. Αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι το τι γίνεται στην Ασία. Έχουμε λοιπόν ε, τις νεοφύης ε, επιχειρήσεις οι οποίες ε, χρειάζονται επιπρόσθετη χρηματοδότηση προκειμένου να αναπτυχθούν γρήγορα. Και συχνά τελικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν ιδέες που να χρηματοδοτούνται και αυτό φυσικά είναι ατυχές γιατί με την έλλειψη χρηματοδότησης στην Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι ιδανικά. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη όθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατοχήρωση αυτού του διαβατηρίου, το οποίο θα προωθεί ακριβώ το επιχειρηματικό κεφάλαιο. Τον Απρίλιο, ωστόσο, του 2016. Μόλις 70 ήταν τα έργα τα οποία είχαν καταθέσει σχετική, σχετική αίτηση. Και νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα τα οποία ενέχει το σύστημα προκειμένου τελικά να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, υπάρχουν προβλήματα καταχώρησης των επιχειρήσεων, καταχώρηση των έργων. Παρουσιάζονται λοιπόν ε, πάρα πολλά εμπόδια σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Άρα, το σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και θα, θα σε πολλές περιπτώσεις να λειτουργεί αντίστροφα. Τι και το θέμα της χρέωσης σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε λοιπόν το όλο σύστημα να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Για να υπάρχει και follow-up ε, χρηματοδότηση, αν χρειαστεί, όπως σας είπα, σε ό,τι αφορά λοιπόν την προοπτική βελτίωση σε τη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιλαμβάνεται αυτό στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αυξηθεί σημαντικά το επιχειρηματικό κεφάλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και η ιδέα είναι να προσελκύονται κεφάλαια και μεγάλοι θεσμικοί επενδυτέ. Τίθεται και το θέμα τη εθνική ε, φορολογία, το οποίο φυσικά την αποτελεί η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Αλλά νομίζω ότι με μικρά μικρά βήματα μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός, προκειμένου αυτές οι πέντε βασικές ε, αρχές να προωθηθούν και να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κεφάλαια αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σβέλλα. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία είναι σημαντικό βήμα για να οριστικοποιήσουμε ένα ακόμη ε, στάδιο της ε, Ένωσης Κεφαλαιογόρων. Μιλούμε για τι εταιρείε επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Το επιχειρηματικό κεφάλαιο είναι σημαντικό ε, χρηματοδοτικό εργαλείο ε, για τι νεοφυεί επιχειρήσει κατά την ίδρυσή του και την πρώτη του επέκταση. Η παροχή εξειδικευμένη χρηματοδότηση, το επιχειρηματικό κεφάλαιο, ε, μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων μπορούν να συμπληρωθούν κενά τα οποία δεν μπορούν να συμπληρωθούν αλλιώ. Αυτή τη στιγμή δυστυχώ η Ευρώπη υπολείπεται άλλων αγορών τα, ε, οι ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι κατακαιρματισμένες, εντοπίζονται σε λίγα κράτη-μέλη και πολλές φορές δεν είναι μεγάλης κλίμακας. Ο αρχικός κανονισμός προσπάθησε να ε, γεφυρώσει αυτά τα κενά δημιουργώντας ε, ευρωπαϊκά σήματα, το, το eu και το EUSEF, προκειμένου να μπορούν τα επιχειρηματικά κεφάλαια να διατίθενται στην αγορά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το EU10 είχε κάποια επιτυχία. 126 ε, τέτοιες εταιρείες έχουν ε, ε, κοινοποιηθεί έως τον προηγούμενο μήνα, αλλά αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Για το EUSEF η πρόοδος ήταν πολύ χαμηλότερη, με μόνο 7 ταμεία να έχουν κοινοποιηθεί μέχρι στιγμής. Βάσει του προγράμματος αυτού λοιπόν και των εξελίξεων αυτών η Κομισιόν αποφάσισε να κάνει την αναθεώρηση των σχετικών κανονισμών και των σχετικών αυτών σημάτων ε, μεγάλη της προτεραιότητα, υψηλή της προτεραιότητα προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση μέσα αυτών των κεφαλαίων των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα ε, προτείνουμε τρεις βασικές αλλαγές προκειμένου να ενισχύσουμε την ανάπτυξη αυτών των ταμείων. Πρώτον, ε, η επιλεξιμότητα των διαχειριστών των ε, ταμείων και η χρήση των EU10 και eu θα περιλαμβάνει πλέον ε, τους διαχειριστές. Με άλλα λόγια, τα περιουσιακά στοιχεία ε, ε εταιριών και ταμείων με περισσότερα, με περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου τα χρήματα αυτά να κατευθύνονται κατευθείαν σε επενδύσεις. Δεύτερον, ε, επεκτείναμε την ικανότητα των ε, ταμείων EU10 προκειμένου να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων. Αυτό θα ενισχύσει την διαφοροποίηση και την ποικιλομορφία προκειμένου να προσελκυθούν περισσότερο, περισσότεροι επενδυτές. Επίσης, μειώσαμε το κόστος απαγορεύοντας τις, τα τέλη και τις χρεώσεις όταν δεν εκτελείται εποπτική λειτουργία. Επίσης, απλουστεύσαμε τις, ε, τους κανόνες καταχώρησης. Οι νέοι κανόνες για τα ταμεία EU10 αποτελούν ε, ένα τμήμα των μέτρων που λαμβάνουμε προκειμένου να ενισχύσουμε την καινοτομία στην Ένωση Κεφαλαιογορών. Μέσω της νομοθετικής διαδικασίας οι νομοθέτες έχουν, έχουν επιβεβαιώσει την δέσμευσή τους προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητοι συμβιβασμοί. Το τελικό κείμενο προσφέρει βεβαιότητα και απλότητα προκειμένου να μπορούν όλα αυτά τα, τα ταμεία να λειτουργούν μέσω των διαχειριστών τους. Επίσης λάβαμε βήματα προκειμένου να ενισχύσουμε τον ρόλο του ΕΣΜΑ προκειμένου να εξασφαλιστούν συνεκτικές και συνεπείς πρακτικές από την πλευρά των εθνικών αρχών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν χαιρετίζει αυτές τις εξελίξεις που θα αναζωογονήσουν τα δύο σήματα EU10 και EU-SEF. Συνάδελφοι, Εγκρίνοντας την πολιτική συμφωνία θα βοηθήσετε την Ευρώπη να ε, προσεγγίσει την, ε, τον στόχο της υψηλής ε, οικονομικής ανάπτυξης με την αξιοποίηση αυτών των εταιριών επιχειρηματικών κεφαλαίων και των Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την εισηγήτρια, του Σκιώδης, αλλά και τον κύριο Γκουαλτιέρη για τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλες οι πλευρές κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων. Ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε, ο κύριο Στόλγεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ένα αδύναμο συμπείο των κεφαλαιοδικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ανεπάρκεια των εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Ίσως είναι η πιο σημαντική ποιοτική διαφορά μεταξύ Τών ε, της αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των ΗΠΑ στις Ηνωμένε Πολιτείε, Αυτές οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου χρηματοδοτούν ε, κυρίως start-up στον τομέα της καινοτομίας. Γι' αυτό δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε μέσω της εισηγήτριας και όλων όσων εργάστηκαν σε αυτό το σχέδιο επειδή μέσω των μέτρων που προτείνονται βελτίνονται οι συνθήκες τόσο ίδρυσης αλλά όσο και ανάπτυξης αυτών των εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Ανοίγει η δυνατότητα να χρηματοδοτούνται startup και για τις ε, μεσές και τις μικρές επιχειρήσεις αλλά και ενισχύεται ο ρόλος των ευρωπαϊκών της Ευρωπαϊκής Αρχής ε, της ΕΣΜΑ. Εγώ θα υπερψηφίσω λοιπόν την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοτσολίνο. Η αναθεώρηση των Γιουβέκα ε, και του ΕΣΕΦ έχουν ε, θετική συνέπεια για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης, για τη δημιουργία πιο σταθερών θέσεων εργασίας και καλύτερων συνθήκων για τις επενδύσεις. Ε, οι εταιρείε επιχειρηματικού κεφαλαίου χρηματοδοτούν ε, κυρίως ε, καινοτόμες εταιρείε πολύ ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν πολύ καλό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και εγώ είμαι μάρτυρας πολλών ε, εμπειριών στη χώρα μου, στην Ιταλία, ε, από επιχειρήσεις που μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν ε, αυτά τα ταμεία. Καταρχήν περιμένουμε σε τέσσερις διαστάσεις. Ε, ε, ουσιαστικά διευρύνουμε το, την κάμα όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, αυτά τα εργαλεία. Έτσι λοιπόν διευρύνουμε την οικονομία κλίμακας για τις επενδύσεις και έχουμε μειώσει το κανονιστικό κόστος που υπάρχει σήμερα. Δεύτερη επιλογή που κάναμε, καταστήσαμε αυτές τις εταιρείε και τα ταμεία ευρωπαϊκά έχουμε δημιουργήσει και απλουστεύσει τις διαδικασίες καταχώρησης σε όλα τα κράτη-μέλη με καλύτερο συντονισμό μέσω της ΕΣΜΑ. Τρίτον, είναι πιο ε, ασφαλή αυτά τα ταμεία και οι εταιρείε ε, γιατί έχουν καλύτερες εγγύσεις ως προς τη διαχείριση. Και τέλος ε, υπάρχει και μία υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για το ΙΟΥΣΕΦ για να μας πούν πώς έχουν ληφθεί υπόψη στους τρόπους επενδύσεων, οι περιβαλλοντικές και οι κοινωνικές πτυχές. Με αυτό το νέο κανονισμό εμείς ενθαρρύνουμε την κοινωνική επιχειρηματικότητα που είναι προηγμένη τεχνολογικά και δίνουμε μεγαλύτερη όθηση στις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, δημιουργούμε ε, μια χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία και δίνουμε περισσότερη προσοχή στο περιβάλλον. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που πετύχαμε και σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Ευχαριστώ κύριος Παπαδημούλης χρειάζεται να ενισχύσουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις την νεανική επιχειρηματικότητα την καινοτομία. η πρόταση της κομισιόν κάνει με καθυστέρηση ένα βήμα μπροστά και η πρόταση του ευρωκοινοβουλίου με τη συμβολή της κυρίας πετικάινεν και των σκιωδών εισηγητών βελτιώνει την πρόταση της κομισιόν. αλλά χρειάζεται να τρέξουμε γρηγορότερα γιατί η απόσταση που χωρίζει τη στήριξη της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων στην ευρώπη σε σύγκριση με άλλες οικονομίες παραμένει μεγάλη. άρα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις να μειώσουμε το κόστος της γραφειοκρατίας περισσότερο να διευκολύνουμε όσους έχουν σπουδαίες ιδέες αλλά δεν έχουν τα κεφάλαια και πρέπει να νοιαστούμε περισσότερο για τις χώρες όπου υποφέρουν περισσότερο όπως η χώρα μου η ελλάδα από την ύφεση και σπουδαία μυαλά μεταναστεύουν στο εξωτερικό γιατί δεν έχει τη δυνατότητα το τραπεζικό σύστημα της χώρας τους να στηρίξει επιχειρηματικές ιδέες. άρα χρειαζόμαστε σε αυτό το θέμα περισσότερα βήματα και περισσότερη ευρώπη. Κύριε Παπαδημούλη, μπλε κάρτα από τον κύριο Κόμπρουν. Σα ευχαριστώ κύριε Παπαδημούλη. Δεν θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι οι κυβερνήσει γενικά είναι ανίκανε γενικά. Δεν είναι οι καλύτεροι δυνατοί άνθρωποι. Γραφειοκράτε που δεν έχουν εμπειρία από την επιχειρηματικότητα. Τι δουλειά έχουν να μπλέκονται σε αγορές, στα χρηματιστήρια. Σίγουρα ο καπιταλισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να βεβαιωθούμε ότι θα αναπτυχθούν οι καινούργιες επιχειρήσεις και με πάσα ειλικρίνεια εγώ ήμουν επιχειρηματής 30 χρόνια τώρα. Αν υπάρχει λοιπόν ένα καλό σχέδιο και αν υπάρχει κανένα καλό έργο, κάποιο θα θέλει να του βάλει χρήματα. Γιατί να σπαταλούμε λοιπόν τα χρήματα των φορολογουμένων Α τα αναλάβει το χρηματιστήριο και οι χρηματοπιστρικέ αγορέ. Ε, Αυτέ είναι νοησίε και σπαταλάμε τα χρήματα των ε, φορολογουμένων. Κύριε Κόμπορν, εσεί που θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν τη Σοβιετική Ένωση, είναι λογικό να θεωρείτε ότι η βοήθεια νέων ανθρώπων να αναπτύξουν νεοφυείς επιχειρήσεις είναι κάτι επικίνδυνο και κακό. Πιστεύετε ίσως σε έναν καπιταλισμό ζούγκλα χωρίς ρυθμίσεις. Διαφωνώ μαζί σας. Δεν συμφωνώ καθόλου όσον αφορά δε τις επικρίσεις για τις κυβερνήσεις μπορεί εσείς να έχετε δίκιο επικρίνοντας την κυβέρνηση της χώρας σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Por favor, silencio. Ο κύριος Μόνο. Μόνο. Monsieur le Commissaire, j'espère que vous prêterez... Πιστεύω ότι θα πρόσεξετε την παρέμβασή μου, κύριε Επιτροπέ. Σα ομολογώ ότι είχαμε βαριέ αμφιβολίε για την αναγκαιότητα που δείχνει η Κομισιόν να αναπτύξει οπωσδήποτε τη, τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών αγορών. Αυτό γίνεται εις βάρος της παραδοσιακής τραπεζικής χρηματοδότησης, εις βάρος της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών. Μία αναθεώρηση του κανονισμού για ε, τον κανονισμό εταιρεών επιχειρηματικού κεφαλαίου και των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θετήθηκε μόλις πριν τέσσερα χρόνια μας φαίνεται κάτι πρόημο. Ε, αυτά τα δύο σήματα χρειάζονται χρόνο ε, για να δείξουν τα αποτελέσματά τους. όμως τώρα η Κομισιόν θεωρεί ότι δεν είναι ε, αρκετά πανευρωπαϊκά αυτά τα σήματα και είναι πολύ μικρά. Και κοιτάξτε, πολλές φορές ε, το μικρό σημαίνει επιτυχία. Μία τέλεια ε, γνώση των κανονιστικών συνθήκων πολλές φορές σημαίνουν ότι θα σημειώσουν κάποια επιτυχία οι διαχειριστές που δραστηριοποιούνται στο τοπικό επίπεδο. Όμως ε, εδώ, ε, καθώς δίνεται αυτό, δίνεται αυτό το σήμα σε διαχειριστές εναλλακτικών ε, οργανισμών σύμφωνα με την οδηγία ΟΔΟΕ. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι οι εταιρείε επιχειρηματικού κεφαλαίου θα βρεθούν πνιγμένα ε, σε διάφορες ε, στρατηγικές ε, που αφορούν τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων. Όμως εμείς θεωρούμε ότι παρά την υποστήριξή μας για τα κεφάλαια κινδύνου θα πόσχουμε στην ψηφοφορία αυτού του κειμένου. Ο κύριε Μονό. Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Κόμπουρν, δέχεστε. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Μάλιστα, ο κύριος Μανώ πολύ γοητευτικό συνήθως. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύω ότι αυτά τα επιχειρηματικά κεφάλαια θα δοθούν σε κάποιες ε, εταιρείε κάπου δεν ξέρω αν έχετε εσεί τέτοιο πράγμα. Εμεί στη Βρετανία δεν έχουμε τέτοιου είδου επιχειρηματικά κεφάλαια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να δοθούν χρήματα σε τέτοιου είδου εταιρείε ει βάρο άλλων εταιρεών που έχουν βρει τα χρήματα μόνε του, γιατί είναι καλό προφανώς αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν ένα πλεονέκτημα, έναν διάλογο που προσπάθησαν ε, μόνοι τους να εξεύρουν τα χρήματα. Προφανώς ο κομμουνισμός έχει ε, επιστρέψει. Ε, εκεί οδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το γεγονός οφείλεται και, και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Ε, η επιχειρηματικότητα ε, έχει καταστραφεί. Εγώ δεν θα ήθελα όμως να δω και τη Γαλλία να καταστρέφεται. Συμφωνείτε μαζί μου σε αυτό. Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα έχετε, όχι ένα λεπτό. Σας το υπενθυμίζω κύριε Μονό. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Κόμπερ, Νομίζω ότι συμφωνούμε σε πολιτικό επίπεδο. Είμαστε και δύο συντηρητικοί, φιλελεύθεροι. Βέβαια, είμαστε αντίθετοι στον κομμουνισμό, στον σοσιαλισμό, σε όλες τις μορφές οικονομικού εξτρεμισμού. Απλώς είμαστε υπέρ του καπιταλισμού και φυσικά είμαστε υπέρ ε, του κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου. Το μόνο πρόβλημα που δεν καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι πριν να υπάρχει υπήρχαν ε, αγορές επιχειρηματικού κινδύνου για χρηματοδοτούν ε, τις νοσίστατες επιχειρήσεις κτλ. Και φυσικά τα κράτη δεν περίμεναν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να λάβουν ε, δράση και να επενδύσουν. Απλώς αυτό ήθελα να πω και γι' αυτό εμείς θα θεωρούμε ότι δεν είναι καλή αυτή η νομοθεσία και θα απόσχουμε από την ψηφοφορία. Κύριε Φερνάντες, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και φυσικά να ευχαριστήσω και τον Ρίκο Σολίνο ε, ως σκιώδη εισηγητή. Ξεκινήσαμε αυτή τη θητεία με μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση στην Ένωση και με σχέδια για να προωθήσουμε την εσωτερική ζήτηση για να βελτιώσουμε την δραστηριότητα και να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και θέλαμε να προωθήσουμε την ε, κεφαλική αγορά. Και εργαστήκαμε πολύ τα τελευταία χρόνια. Είχαμε το νέο κανονισμό ε, για ε, τα νομισματικά ταμεία, την ε, οδηγία προσπέκτους. Είχαμε μια τελευταία συμφωνία στον τριμερή διάλογο για να έχουμε πρότυπη τιτλοποίηση σε επίπεδο Ένωση. και ο κανονισμός που συζητάμε σήμερα και που θα ψηφίσουμε νομίζω ότι οδεύει στην ε, ίδια γραμμή να οικοδομηθεί αυτή η εσωτερική αγορά κεφαλαίων μέσω της διευκόλυσης της δημιουργίας εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου και ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Είναι μεγάλη η πρόταση αυτή. Η δική μου ομάδα εργάστηκε σκληρά και σημειώσαμε πρόοδο σε ό,τι αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο της ΕΣΜΑ και στο να διευκολύνουμε τις επενδύσεις σε μικρότερες επιχειρήσεις εισάγοντας και ανάλυση περιβαλλοντική, προκειμένου να σεβόμαστε και τη Συμφωνία του Παρισιού. Και θεωρώ ότι πήραμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Τώρα, πέρα από όλα όσα κάναμε, όπως είπε και ο συνάδελφος Παπαδημούλης, μας μένουν ακόμη πολλά να κάνουμε, γιατί οι μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν σημαντικές προκλήσεις για να μπορούν να συμμετέχουν στην ενιαία αγορά. Υπάρχουν πολλά διοικητικά προβλήματα, κανονιστικά προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε ένα μέρος αυτών των μεταρρυθμίσεων ουσιαστικά απευθύνονται σε μεσαίες επιχειρήσεις που ήδη συμμετέχουν στις κεφαλαϊκές αγορές και θα πρέπει να σκεφτούμε και απευθύνομαι στην Κομισιόν πώς μπορούμε πράγματι να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις και όχι μόνο για τις μεσαίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που θα αναλάβω την Προεδρία της Ολομέλειας σήμερα το απόγευμα και θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Άνεμανς από το ΙΕΝΕΦ. Στον κύριο Άνεμανς. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, ακούσαμε σήμερα το πρωί από τον Ζανκλοντ ε, Γιούγκερ, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεφαλαία Αγορά να πάει σε υψηλότερη ταχύτητα. Και μετά από αυτά που ακούσαμε στην, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ό,τι αφορά το Brexit με τόσο πολλούς ε, εργαζόμενους στις κεφαλαίες και στις, ε, το City του Λονδίνου αποτελεί ένα από τα ε, σημαντικότερα, από τα σημαντικότερα μέρη και θεωρούμε ότι είναι μεγάλη πρόκληση και θα πρέπει να είναι σωστή η απάντηση στα υπερβολικά φιλοδόξα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημά μας λοιπόν που αντιμετωπίζουμε με την έκθεση αυτή. Και επίσης θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να είναι η ΕΣΜΑ, αλλά τα κράτη-μέλη αυτά που θα αναλάβουν ε, την πρωτοκαθήδρια για να υπάρξει η ενοποίηση της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης που είναι κατά της ε, Ευρωπαϊκή ε, Υπήρου, γιατί η ομόνια και η ενότητα βγαίνει από την διαφορετικότητα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Σαντ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρότασή μα εδώ πέρα ε, προσπαθεί να καλύψει ένα βασικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των νεοφιών επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν η χρηματοδότηση αυτή να, ε, να κινητοποιείται από οτισείς και από διάφορους τέτοιους δημοσιολογητές. Αλλά θα πρέπει να υποτιμούμε και τις δυσκολίες που υπάρχουν ε, αυτοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πυρός σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα και την, ε, τον καθορισμό της νομοθεσίας. Θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, να είναι καινοτόμοι και να προσαρμόζονται στις συνθήκες που απαντούν. Η αποτελεσματική λοιπόν νομοθεσία θα πρέπει να είναι ελαφριά γιατί οι νεοσύστατες ε, επιχειρήσεις ε, κυρίως επικεντρώνονται και στο ψηφιακό περιεχόμενο και στον τομέα της ψυχαγωγίας. Ε, θα πρέπει να προαχθούν και επιχειρήσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών, των περιβαλλοντικών ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Χρειάζεται λοιπόν διαφοροποίηση και θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των επιχειρηματικών κεφάλαιων και των αντίστοιχων τμήματων των πανεπιστημίων. Χρειάζονται λοιπόν ιδιαίτερα προγράμματα για τις περιφερειακές και τις νησιωτικές περιοχές για να αναπτυχθεί το δυναμικό των μικρών επιχειρήσεων το οποίο απειλείται από την έλλειψη επιχειρηματικού κεφαλαίου σε αυτές τις περιοχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φροντζούλικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρά το γεγονό ότι αποτελεί θεμέλιο του Civil Action Plan, του σχεδίου δράσης, ε, τα, τα μη επιχειρηματικ... κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τα, οι εταιρείε ε, επιχειρηματικών κεφαλαίων περιορίζονται σε λίγα κράτη-μέλη μόνο. Γι' αυτό και χαιρετίζω τις αλλαγές που προτείνονται και προβλέπονται στην έκθεση και νομίζω ότι εκεί περιγράφονται μέτρα τα οποία αποσκοπούν στο να ενισχυθούν τα επιχειρηματικά κεφάλαια και να προωθηθούν τα δύο συστήματα χρηματοδότησης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά, να βελτιωθεί η πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων, όλων των μεγεθών στη χρηματοδότηση σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, Ιδίω η πρόταση για μείωση του ορίου για τις εταιρείε επιχειρηματικών κεφαλαίων σε 50.000 ευρώ είναι πολύ θετική καθώς αυτό θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και θα διευρύνει τις επενδυτικές δυνατότητες. Από την άλλη πλευρά, η αυστηρότερη επαγρύπνηση και παρακολούθηση ε, μέσω του ρόλου που αποδίδεται στον ΕΣΜΑ θα αποσβέσει κινδύνους, θα απορροφήσει κινδύνους για τις χρηματαγορές και θα διευκολύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Ευχαριστώ κύριε Φουρτσουλικά. Περνάμε τώρα στο Κατζιάι. Ο κύριος Καπούτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ στο πλαίσιο της στρατηγικής οικοδόμησης της ε, νέας ε, αγορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλει να υποστηρίξει τις εταιρείε επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Το επιχειρηματικό κεφάλαιο αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις νέες και καινοτόμες και μικρές επιχειρήσεις. Τα δεδομένα του 2015 και 2016 φαίνονται ενθαρρυντικά, όμως τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του κανονισμού EUVK μόνο το 25% του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Κεφαλαίου ε, συλλέχθηκε εκτός των κρατών ε, μελών ε, καταγωγής. Ε, η διεύρυνση του αριθμού των επενδύσεων ε, είναι δυνατή βελτιώνοντας τη ροή των εναλλακτικών επενδύσεων και ουσιαστικά ε, επενδύοντας και στο ταλέντο τόσων νέων επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καπούτο. Ο κύριος Μαριάς. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, οι τράπεζες δεν έχουν συνέλθει από την οικονομική κρίση και αυτό που κάνουν βεβαίως είναι να μην δίνουν κεφάλαια επενδυτικά στις μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. έτσι είναι αναγκαία να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά κεφαλαίου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης και σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει μια διευκόλυνση για την ίδρυση εταιριών επιχειρηματικού κινδύνου και ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας για να στηριχθούν οι νεοφυεί επιχειρήσει σε όλες τις χώρες και κυρίως στην ελλάδα όπου όμω, στην ελλάδα θα πρέπει να επισημάνω ότι η τράπεζα τη Ελλάδο, η οποία συμμετέχει στην ποσοτική χαλάρωση έχει δαπανίσει 42,5 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ θα έπρεπε μέρος αυτών των χρημάτων να έχει βρει τρόπο να μπορέσουν να δαπανηθούν υπέρ εταιρικών ε, διαδικασιών δηλαδή υπέρ εταιρικών ομολόγων και κυρίως μέσα από αυτή τη διαδικασία να στηριχθούν και οι νεοφυείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη να έχουν χρηματοδότηση προκειμένου να υπάρξει επιτέλους ανάπτυξη στην ελλάδα η οποία έχει χτυπηθεί από τη σκληρή πολιτική της τρόικας και αυτή τη στιγμή έχουμε εκατομμύρια ανέργους. ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ε, και με αυτό ολοκληρώνουμε τη διαδικασία Catch Επομένως, θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον Επίτροπο Βέλα για να μας πει τη γνώμη της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, για τα σχόλια και για την υποστήριξη που πολλοί από εσάς εκφράσατε για τη συμφωνία αυτή. Όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το θέμα αυτό είναι ε, επίγουσας ανάγκης για την ε, ε, δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαιογορών και σας ευχαριστούμε για την επικοδομητική σας στάση. Φαίνεται ότι χάρη σε αυτήν τη στάση θα συνεχίσουμε να κάνουμε γρήγορη πρόοδο. Ε, για την αναζωογόνηση των σημάτων EU10 και EUSEF, ε, η αναζωογόνηση μάλλον, θα δημιουργήσει περισσότερες ε, πηγές χρηματοδότησης για την υποστήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεών μας. Αποτελεί ένα βήμα προς την οικονομία του μέλλοντος. Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον την, την εισηγήτρια, τους σκιώδεις εισηγητές και τον κύριο Γκουαλτιέρη για το έργο τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, κύριε Επίτροπε. Η εισηγήτρια τώρα, η κυρία Πιετικάινεν, δύο λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την επικοδομητική της στάση κατά τη συνεργασία που είχαμε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ε, και για το γεγονός ότι καταφέραμε να έρθουμε σε συμφωνία. Ωστόσο, θα ήθελα να σας πω δύο ακόμη πράγματα. Πρώτον, Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια βήματα όσον αφορά το EU που είναι το αρχικό κεφάλαιο και η δυνατότητα ε, επένδυσης ε, με μεγαλύτερη ευελιξία. Πρέπει αυτό να το δούμε στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον όταν θα γίνει η αναθεώρηση του κανονισμού. Τι είναι το σημαντικότερο. Τώρα που η Κομισιόν θα κάνει την αναθεώρηση του ΕΣΜΑ, ελπίζω να αναλάβετε τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να εξασφαλίσετε ε, με διαφανή τρόπο την ε, πανευρωπαϊκή μεταχείριση των ε, ταμείων EU10 προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος τους γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι πραγματικά ε, η λιδία λήθος για την δημιουργία μιας εύρυθμης λειτουργίας των, της, της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών και ενός συστήματος